έκθεση του 2005 για την Τουρκία. Και ευθύ εμέσω ο λόγο στην κυρία Χένι Πλέσσερ για το Συμβούλιο. Για την Τουρκία. Too many debates. Η μία συζήτηση διδέχεται την άλλη. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, Αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία έχει στρατηγική σημασία και έχουμε μακρά ιστορία ε, ευρύτατη συνεργασία. Έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, αλλά παράλληλα έχουμε και πολλές κοινέ προκλήσεις. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από την κρίση του μεταναστευτικού προβλήματος και ο πρόεδρος Τούσκ το ανέφερε προηγουμένως. Οι διαπραγματεύσει ε, για την ένταξη συνεχίζονται, όπω ξέρετε. Ανοίξαμε το τελευταίο κεφάλαιο το 17 το Δεκέμβριο και ε, το 33 ε, σκοπεύουμε να το ανοίξουμε με την Τουρκία κατά τους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο των κανόνων ένταξης με ομοφωνία σύμφωνα με τις βασικές προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργούμε, χωρίς να ελαφρύνουμε τις προϋποθέσεις. Από την έκθεση της Επιτροπής είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς του κεκτημένου και αυτό είναι πολύ θετικό νέο. Παράλληλα είναι εξίσου σαφές ότι πολλές τρέχουσες εξελίξεις και ανησυχητικά συμβάντα στην Τουρκία μας δημιουργούν ε, λόγω ανησυχίας. Η Τουρκία θα πρέπει να επανορθώσει σημαντικές υστερήσεις, ιδίως στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Συμβούλιο ζητά από την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβει επίγοντα μέτρα για να αντιστρέψει τα μέτρα υπονόμευσης ε, του δικαστικού σώματος ε, και να βελτιώσει ε, την κατάσταση στα θέματα του δικαιώματος του συνέρχεστε και του δικαιώματος έκφρασης. Είναι σημαντικά και ιδιαίτερα επίγοντα θέματα τα οποία καταγράφονται και στο δικό σας ψήφισμα. Όπως επανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο, αναμένουμε από την Τουρκία ότι θα τηρήσει τα ύψιστα πρότυπα τα οποία έχουμε. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Τουρκία επαναλαμβάνουμε αυτές τις ανησυχίες μας σε κάθε ευκαιρία και επανειλημμένα ζητάμε την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για να σταματήσει η βία στη νοτιοανατολική Τουρκία και να βρεθεί μια επίγουσα λύση στο πρόβλημα με, στο κουρδικό ζήτημα. Θέλω να επαναλάβω ε, ε, ότι χαιρετίζουμε την δέσμευση των δύο μερών για την ε, επίλυση του προβλήματος με την Κύπρο. Υποστηρίζουμε την Κύπρο στην προσπάθεια που κάνει και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Χάν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Κάτι Πύρη για την υψηλή ποιότητα της έκθεσης που συζητάμε σήμερα. Ασχολείται με τα βασικά ζητήματα των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά συμφωνεί με τα ευρήματα της Επιτροπής στο πακέτο για την διεύρυνση το και με την έκθεση για την Τουρκία στα πλαίσια της ε, κρίσης των προσφύγων και των μεταναστών και την πολιτική κατάσταση της περιοχής και επειδή έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα ως Ένωση με την Τουρκία είναι ζωτικό να αναζωογονήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με αυτόν τον στρατηγικό εταίρο. Φυσικά, οι σχέσεις μας πρόσφατα εστιάστηκαν στις προκλήσεις του μεταναστευτικού αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να ασχολούνται και με πολλά άλλα θέματα, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό αυτής της σχέσης. Η πιο η επανενεργοποιημένη διαδικασία ένταξης είναι ο πυρήνας ε, της κοινή μας προσπάθειας. Ε, το άνοιγμα κεφαλαίων ελπίζουμε να οδηγήσει σε συγκεκριμένη πρόοδο στην Τουρκία. Με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία τη 18 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εκπονεί μια πρόταση προ το Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ε, οι ενταξιακές για θέματα οικονομικά και δημοσιονομικά. Είμαστε επίσης σε φάση προετοιμασίας ε, ανοίγματο νέων κεφαλαίων για το δικαστικό τομέα, θεμελιώδη δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και ασφάλεια. Τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς να προκαταλαμβάνουμε τη θέση των κρατών μελών και σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή ενθαρρύνεται από την πρόοδο στις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού και προσβλέπουμε σε ε, σύντομη και επιτυχή κατάληξή τους και βασιζόμεθα στην μόνιμη και διαρκή συμβολή της Τουρκίας στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας τέτοιας συνολικής λύσης. Θα ήταν πολύ καλό για την ασφάλεια και για την, ε, για την Ευρώπη, συγγνώμη, και για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή να υπάρξει μια τέτοια λύση και θα συνέβαλε σε μια μεγάλη προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ για την ισχυρή βοήθειά σας για διαρθρωμένο διάλογο υψηλότερου επίπεδου. Ο πρόσφατος πολιτικός και ενεργειακός διάλογος κατέδειξαν ότι είναι επιτυχημένες μορφές για να προχωρήσουμε το κοινό μας θεματολόγιο με την Τουρκία. Και ένας διάλογος υψηλού επίπεδου στις 25 και 26 Απριλίου θα βοηθήσει να αυξηθεί η συνεργασία στον επιχειρηματικό τομέα και θα επιτρέψουν συζητήσεις για μακροοικονομικά θέματα, οικονομική πολιτική και δυνατότητες επενδύσεων. Όπως είπαμε και το πρωί, η σφαιρική προσπάθεια, συνεργασία μας με την Τουρκία για το μεταναστευτικό έχει δώσει πρώτα αποτελέσματα για να επιτύχουμε το στόχο μας να σταματήσει η, η παράτυπη μετανάστευση από την Τουρκία στην Ένωση και να σταματήσει αυτή ε, η προσπάθεια που κάνουν οι μετανάστες και πρόσφυγες που σημαίνει ότι κινδυνεύουν τη ζωή τους. Θέλουμε να βασιζόμεθα στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Τουρκία. Και έχουμε ανησυχίες γι' αυτό. Και οι ανησυχίες μας οξύνθηκαν λόγω προσφάτων εξελίξεων, όπως αυτές που αφορούν την ελευθερία έκφρασης ε, πανεπιστημιακών ή δημοσιογράφων και αποφάσεις για ιδιωτικά ΜΜΕ. Έχουμε καλέσει την τουρκική κυβέρνηση να επανέλθει σε μεταρρυθμίσεις για να φτάσει σε ευρωπαϊκού επίπεδου επίπεδα προδιαγραφές μάλλον σε αυτούς τους τομείς. Και ελπίζουμε ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 θα συμβάλλουν ουσιοδός στο να ανανεωθεί η δέσμευση της Τουρκίας για μεταρρύθμιση σε αυτούς τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης συνεχίζει να εκφράζει τις ανησυχίες της για τη σοβαρή κατάσταση στην νότια ανατολική Τουρκία. Χρειάζεται γνήσιος πολιτικός διάλογος στα πλαίσια της διαδικασίας διευθέτησης του Κουρδικού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ειρηνική και βιώσιμη λύση. Και η Ένωση είναι διατεθειμένη να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Καταλήγοντας, η Επιτροπή έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία θα βοηθήσει να επιλύσουμε τη μεταναστευτική κρίση και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας σε πολλούς άλλους τομείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε στου αγορητέ από τι πολιτικέ ομάδε. Η κυρία Πύρη από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν παρόμοιε προκλήσει. Σκεφτείτε την κρίση των προσφύγων, την τρομοκρατική απειλή και τον πόλεμο στη Συρία που δημιουργεί αστάθεια. Ένα πράγμα έχει καταστεί σαφέ μετά από τι κοινέ αυτέ προκλήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία χρειάζονται μια την άλλη για να αντιμετωπίσουν με κοινέ λύσει τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο, και αυτό θέλω να το τονίσω, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να μην βλέπουμε τι εσωτερικέ εξελίξει στη χώρα. Η Τουρκία πρέπει να σταθεροποιηθεί και πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική, εάν θέλουμε να είναι ένα στρατηγικό εταίρο με τον οποίο να μπορούμε να συνεργαστούμε. Το να διασυνδέσουμε την συνεργασία μα για την μετανάστευση με τη διαδικασία προσχώρηση δεν είναι δίκαιο ούτε σωστό. Δεν πρέπει να επιταχυνθούν οι ομιλίε πρωτού γίνουν μεταρρυθμίσει. δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό παρεδό δούνε για να γίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να δούμε και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο τουρκικός πληθυσμός ήδη έχει υποδεχτεί 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν ίσως να μάθουν μαθήματα από τη φιλοξενία που έχουν δείξει οι Τούρκοι. Όμως ταυτόχρονα η Τουρκία φτάνει στα ωριά της. Και επιτέλους πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πλώσει χείρα και να προσφέρει ε, μεγάλα μεγάλη εμβέλεια προγράμματα επανεγκατάσταση των προσφύγων προ τι ευρωπαϊκέ χώρες. Αυτή είναι πραγματική κατανομή του άρθρου και αυτή είναι πραγματική συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλέ ευκαιρίε που μπορούμε να σε επέτρεπε να συνεργαστούμε, αλλά τι χάσαμε. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να έχουμε εντατικότερο και ειλικρινέστερο διάλογο με πραγματικέ μέρημνε που δεν θα πρέπει να τι ε, λαμβάνουμε ως προσβολέ κατάσταση στα νοτιοανατολικά τη χώρα Ανησυχεί ιδιαίτερω αυτό το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει η ειρηνευτική διαδικασία να ε, αποκατασταθεί καθώς δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για το κουρδικό. Η σημερινή κατάσταση, η τρέχουσα κατάσταση του status quo είναι απαράδεκτη. Δεν θέλουμε να υπάρξει επιστροφή στη βία από το ΠΚΚ, ούτε να υπάρξουν επιθέσει κατά των δυναμένων ασφαλεία και των ε, ε, πληθυσμών, των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιτρομοκά από την κυβέρνηση, ταυτόχρονα τονίζουμε ότι πρέπει να είναι αναλογικά και ε, να συνάδουν με το διεθνέ δίκαιο. 400.000 πολίτε έπρεπε να εκτοπιστούν εσωτερικώ λόγω των δύο επεισοδίων και είναι πολλές ε, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας ε, σε πολλές χορτικές πόλεις που έχουν ε, διαταράξει τελείως την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Θέλουμε μια Τουρκία όπου οι δημοσιογράφοι να μην φυλακίζονται γιατί κάνουν τη δουλειά τους και να μην λογοκρίνονται, να μην αυτολογοκρίνονται ενστικτοδός. Θα πρέπει οι πανεπιστημιακοί να μην χάνουν τις δουλειές τους και να μην μπαίνουν στη φυλακή απλώς επειδή εξέφρασαν ελεύθερα τις απόψεις τους. Επιτέλους η Τουρκία πρέπει να επιστρέψει στην οδό που οι δικαστές δεν θα ε, δέχονται οδηγίε ότι πρέπει να αποφασίσουν και να μην λαμβάνουν αποφάσει ε, από φόβο μήπω μετατοπιστούν ή απολυθούν σε μια δημοκρατική Τουρκία που αυτή θέλουμε, τέτοιου είδου ε, συνθήκε επιζητούμε. Πρέπει να επιστρέψει στην οδό των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για στενοτρή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και του συναδέλφου συνεισηγητέ για την καλή συνεργασία που είχαμε και Νομίζω ότι με αυτό το ψήφισμα μπορούμε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πύρη. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Κυρία Πύρη, ακούστε με. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Ο κύριο Κριστοφόρου. Παρακαλώ. Κύριε Κριστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε. Αναμένω από την εισηγήτρια τη έκθεση να μα πει εδώ ξεκάθαρα εάν αισθάνεται ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν προχωράει η ενταξιακή πορεία τη Τουρκία γιατί η τουρκία ουσιαστικά αρνείται να εφαρμόσει και να υλοποιήσει όχι τώρα που είναι το προσφυγικό αλλά εδώ και χρόνια τα προαπαιτούμενα προ την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θέλει κατά χάριν ουσιαστικά είσοδο και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά με όλε τι άλλε χώρε και αυτέ που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτέ που είναι υποψήφιε για ένταξη υποχρεωτικά πληρούν όλα τα κριτήρια. Και ένα τελευταίο, είναι δυνατόν η εισηγήτρια να αναφέρει ότι πρέπει να γίνει ακόμα και σήμερα άνοιγμα των κεφαλαίων χωρί η τουρκία να τηρήσει τα προαπαιτούμενα. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση συνάδελφε. Είναι σαφές Θα ήταν ε, αρκετά σκληρό να επερευνούν τι ευθύνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι οι διαδικασίε δεν επιταχύνονται. Τι ευθύνε τι έχει η τουρκική κυβέρνηση, για μένα είναι σαφέ. Και βεβαίω αυτή είναι και η ουσία τη διαδικασία. Πρέπει να αξιολογήσουμε την Τουρκία όπω αξιολογήσαμε άλλε υποψήφιε χώρε. Και εδώ πρέπει να πω ότι ε, υπήρξαν πολιτικέ διαφορέ ε, που κάποιοι τις εκμεταλλεύτηκαν στην Ευρώπη με πολιτικά παιχνίδια και δεν έχει τύχει πάντοτε δικές μεταχείρισης ε, η Τουρκία όπως άλλες χώρες. Ευχαριστούμε κυρία Ζόμερ για δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Κάτι Πύρη για τη συνεργασία και τους κοιόδης των άλλων πολιτικών ομάδων. Συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό με βάση το ψήφισμα της περσινής χρονιάς να εργαστούμε και το επιτύχαμε. Και αυτό απλοποίησε τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω κάτι. Γιατί τώρα, τελευταία στιγμή, δεν τηρήσω όλα τα συμφωνημένα. Όταν βλέπω ότι οι σοσιαλιστές συμφωνούν με, τη, με τον κατάλογο ψηφοφοριών του ΕΛΚ. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πιέστε το ΕΛΚ. Δεν θα πιεστεί το ΕΛΚ από καμία άλλη πολιτική ομάδα, ούτε από το κύμα των προσφύγων. Το καθήκον μας είναι μέσω του ψηφίσματος να αποτιμήσουμε την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία για να δούμε αν προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να το μπλέξουμε με την προσφυγική κρίση όσο δύσκολη και αν είναι. Για μας είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις έναντι της Τουρκίας. Αυτό ισχύει για τη φιλελευθερωπή των θεωρήσεων, για την οποία πρέπει ε, να ισχύσουν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις και το άνοιγμα κεφαλαίων αυτονόητα πρέπει να συνεχίσει να συνδέεται με την εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων από την Τουρκία. Αλλά απέχει πολύ η χώρα από αυτό. Η ελευθερία του τύπου, της έκφρασης των διαδηλώσεων, βασικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ε, κουρδικό θέμα, βία στην ε, νοτιοανατολική Τουρκία. Βήματα προς τα πίσω. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς ε, γείτονες της Τουρκίας, αν θέλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας, τότε πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε ένας με τον άλλον και να διαπραγματευτούμε. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν η Τουρκία αποφασίσει να οδεύσει την Ευρωπαϊκή Οδό. Και τα κεφάλαια που σχετίζονται με την Δημοκρατία της Κύπρου ποτέ δεν θα ανοίξουν αν δεν επιληθεί το Κυπριακό. Η Τουρκία πρέπει να γίνει πιο επικοδομητική. Πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να καταλάβει ότι μόνο με την ε, ε, βάση των ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να υπάρξει επανένωση και είναι και προς το συμφέρον της Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος εκ μέρους της Ομάδας των Ευρωπαίων και Ευχαριστώ. Διαβάζοντας την έκθεση αυτή, ε, βλέπουμε ότι ε, επικρίνεται η αυταρχική στάση του Προέδρου Ερντογάν. Είχα αναφέρει και στο παρελθόν την αγανάκτησή μου έναντι του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τους δημοσιογράφους και έναντι της έλλειψης ελευθερίας του τύπου και ελευθερίας της έκφρασης. Και σε πρόσφατη έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι σε πολύ χαμηλή θέση ε, ε, μεταξύ των ε, χωρών διεθνώς. Αναφέρετε τις ανησυχίες σας, αναφέρετε ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν. Το ζητάτε μένα, αλλά τελικά τι επιτύχατε, τίποτα δεν έχετε επιτύχει. Η νοτιοανατολική Τουρκία παραμένει μια ζώνη εμπόλεμη και η Τουρκία παίζει ένα διπλό παιχνίδι στην, στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους, στο ρόλο που παίζει ε, εναντί των ξένων μαχητών και για τα χρήματα τα οποία πρέπει να φτάνουν στην Συρία και ε, εναντί των Κούρδων μαχητών. Ο κύριος Λάμστορφ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, Είπατε ότι θα, προκύψουν, θα προκύψουν πλεονεκτήματα από την ενισχυμένη συνεργασία με την Τουρκία. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν είμαστε σίγουροι εάν αυτά τα πλεονεκτήματα ε, θα τα επιτύχουμε στα πλαίσια μιας διαδικασίας ένταξης. Γιατί αυτή η διαδικασία έχει περιγραφεί σαν να είναι σε κατάσταση ζόμπι. Στην ε, ουσία έχει πεθάνει. Κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά. Κανείς δεν πιστεύει ότι μια μέρα θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Αυτό που χρειαζόμαστε αντί για αυτό είναι μια σχέση που να βασίζεται σε σεβασμό για την Τουρκία και ρεαλισμό και μια θετική ατζέντα. Υπάρχουν πολλοί τομεί για του οποίου μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Τουρκία και πολλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το προσφυγικό, ενεργειακή συνεργασία, πολιτιστικέ ανταλλαγέ, επαφή μεταξύ των ανθρώπων, τουρισμό, εμπόριο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτό το σημαντικό εταίρο. Αλλά πρέπει να σεβόμεθα ο ένας τον άλλον. Εάν όμως εδώ λέτε ότι κάνετε μια πρόταση για να ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια χωρίς αυτό να προκαταλαμβάνει τη θέση κάποιων κρατών μελών. Και παράλληλα ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει ομοφωνία των κρατών μελών δεν μπορεί να ανοίξουν τα κεφάλαια. Είναι σαφές λοιπόν των προτέρων ότι γίνονται απεγνωσμένε προσπάθειε να διατηρηθεί εν ζωή μια αποτυχημένη διαδικασία. Δεν υπάρχει το αναγκαίο θάρρο για να δημιουργήσουμε νέα βάση για καλέ σχέσει με την Τουρκία. Από τότε που διαπραγματευόμαστε την Τουρκία, είναι 11 χρόνια τώρα. Οι σχέσει μεταξύ τη χώρα και τη Ένωση όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί, έχουν επιδεινωθεί. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι, θα έλεγα, και δηλητηριασμένε. Δείτε πώς συμπεριφέρεται ο πρόεδρος της Τουρκίας έναντι του Γιάνν Ντόμερμαν ενός Γερμανού κομικού. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Αυτά δείχνουν ότι δεν σέβεται την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Να έχουμε το θάρρος να βαδίσουμε ένα νέο δρόμο. Να συνεργαστούμε με την Τουρκία για να φτιάξουμε ένα θετικό θεματολόγιο με σεβασμό, αλλά ας αφήσουμε αυτά περί ένταξη. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό κύριο Χατζηγεωργίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια την Κατυπήρη για την άψογη και παραγωγική συνεργασία της καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Νομίζω ταυτόχρονα ότι η κατάσταση στην Τουρκία υπερκερά κατά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε εδώ για την έκθεση. Μια έκθεση που εν πολλής αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Στην νοτιοανατολική Τουρκία υπάρχουν ήδη περίπου 300.000 εκτοπιστέντες μεγάλο μέρος της πόλης σουρ έχει πλήρως εγκαταληφθεί. μεγάλο μέρος της έχει δημευθεί απαλωτριωθεί. ουσιαστικά δηλαδή πήραν τις περιουσίες 60.000 ανθρώπων. ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι διώκονται απλά και μόνο διότι μίλησαν ελεύθερα. στις 22 απριλίου σε μια εβδομάδα από τώρα γίνεται δίκη αυτών των ανθρώπων στην κωνσταντινούπολη και έχω ήδη πάρει έκκληση από τους κατηγορούμενους όπως μέλη του κοινοβουλίου παραστούν και παρακολουθήσουν τη δίκη ως παρατηρητές. Καλούμε την Τουρκία να αρχίσει άμεσα διάλογο για επίλυση του Κουρδικού και να πάυσει να διώκει ελεύθερη έκφραση. Η απάλληψη και διαγραφή του ΠΚΚ από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει. Η έκθεση περιέχει πολύ θετικέ αναφορέ για το Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένη αναφορά ότι η λύση θα αποτελεί μετεξέλιξη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μέχρι στιγμή όμω περιέχει έμμεσε έστω αναφορέ για άνοιγμα κεφαλαίων πράγμα με το οποίο διαφωνούμε αφού η τουρκία δεν έχει υλοποιήσει υποχρεώσει που ανέλαβε. στο κυπριακό ενώ είναι καλοδεχούμενε θετικέ αναφορέ εκ μέρου τούρκων αξιωματούχων είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξη οι αναφορέ αυτέ. δέκα δευτερόλεπτα κύριε πρόεδρε. αναμένουμε άμεσα κατάθεση χάρτη για το εδαφικό πράγμα που θα διευκολύνει και την επίλυση του περιουσιακού. Πιστεύω πως η Τουρκία, δώστε μου πέντε δευτερόλεπτα, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και στόχος δικός μας είναι να παράσχουμε κάθε βοήθεια στον τουρκικό λαό. Ευχαριστώ. Λυπάμαι, ένα μισή λεπτό είχατε όλο και όλο. Η κυρία Βαλερό για ένα μισή λεπτό από την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θεωρώ ότι οι εξελίξεις στην Τουρκία δεν είναι οι... αυτές που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε εμείς. Δεν ακολουθεί το σωστό δρόμο. Η ελευθερία τύπου έκφραση στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνουν σεβαστά στην Τουρκία. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιθυμήσει ο δρόμος της Τουρκίας να πήγαινε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε επίσης να υπάρξει ειρήνευση με τους Κούρδους, αλλά ούτε και αυτό έχει γίνει πραγματικότητα. Τίποτα τελικά από ό,τι ευχόμαστε δεν έχει πραγματοποιηθεί όλα πηγαίνουν αντίθετα από την κατεύθυνση που θα θέλαμε. Όλοι οι δημοκράτες στην Τουρκία, όλοι αυτοί που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν. Το ψήφισμα φέτος επικρίνει την κατάσταση της Τουρκίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και ζητά και τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις βίες ενέργειες για να προωθήσουν την ειρήνη. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική διαπραγμάτευση χρειαζόμαστε ένα πραγματικό συνομιλητή. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των συνομιλητών από την πλευρά των Κούρδων είναι στη φυλακή. Ο Ετσαλάν βρίσκεται σε απομόνωση στη φυλακή. Δεν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αλληλογραφία, δεν έχει επαφή με κανένα. Ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να δώσει τα μηνύματα στους ε, δικούς του. Εμείς λοιπόν ως πράσινοι θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτή η βία φυλάξη του Ατζαλάν. Έχει το λόγο τώρα. Ο κύριος Κάρδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της Τουρκίας καταδεικνύει μέχρι πού θέλει να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα των νεοαπικιακών της φιλοδοξιών. Καταπατά τα θέματα της δημοκρατίας, των της ελευθερίας του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη δράση της ενώ τα διαδηλώνει σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε φτάσει το, την κορύφωση της υποκρισίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ουσιαστικά δώσει λεφτά για να πληρώσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει μια ολέτρια πολιτική ασύλου. Το ότι η Τουρκία ακόμα και ενδέχεται να, ξεκινήσουν, να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με την Ευρώπη, αυτό καταδεικνύει πως εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα απολύτως. Την τελευταία εβδομάδα οι Ολλανδοί απέριψαν την διεύρυνση της Ευρώπης στο δημοψήφισμα για την Ουκρανία και η υποστήριξη για τον Brexit, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αυξάνεται. Αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί Δανείοι θα κάνουν το ίδιο. Όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που περνάμε μια πραγματική κρίση στην Ευρωζώνη, στην ζώνη του Σέγγεν και έχουμε ένα πρόβλημα με τη μετανάστευση. Η περαιτέρω διεύνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια απειλή προ τη χώρα μου, κυρία Πρόεδρε. Γι' αυτό ο μόνο τρόπο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη Μεγάλη Βρετανία είναι να φύγουμε στι 23 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και μισό ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση είναι ένα αριστούργημα υποκρισίας. Θέλει να θέλουμε να κρύψουμε τα τεκμηριωμένα στοιχεία που υπάρχουν και που αντιτίθεται στην ε, πορεία ένταξης της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της έμφασης και των επένων για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποτίθεται ότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο. Όμω η έκθεση δεν λέει πώς Ποιες φύσεις είναι οι διαδικασίες αυτές φιλοξενίας και ποιες είναι οι πρακτικές μαζικών ε, αποθήσεων που καταγγέλλονται μάλιστα αυτή τη στιγμή από την Διεθνή Αμνηστία. Ένα ερώτημα λοιπόν τίθεται. Η Τουρκία θα πρέπει να θεωρηθεί ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες. Και άλλο ερώτημα. Αυτή η αρχή του περιορισμού που ένα σωρό φορέ έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε όσου στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία έθεταν ε, τα προβλήματα για την ζωέ ε, και την ε, εισβολή των παρανόμων για την Τουρκία δεν ισχύει. Το γεγονός ότι στην Τουρκία εφαρμόζεται μαζικά η αρχή της απόθεσης δεν ισχύει για την Τουρκία. Είναι μια βασική αντίφαση που δείχνει πόσο στρεβλή είναι αυτή η υπέροχη ιδέα για την Τουρκία. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να απορρίψουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων και να ζητήσουμε την επαλήθευση και τον έλεγχο για την πραγματική δέσμευση της Τουρκίας απέναντι στους ξένους μαχητές και να επαληθεύσουμε τις σχέσεις της Τουρκίας με τον ΙΣΥΛ. Βόιτ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέτω στον εαυτό μου το ερώτημα γιατί καταφέρνει η Τουρκία να εκβιάζει με τον τρόπο αυτό την ε, Ευρώπη. Εσείς έχετε ένα κατάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έπρεπε να εκπληρώσει η Τουρκία. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Η Τουρκία παραβιάζει και βεβηλώνει τις χριστιανικές εκκλησίες κατάσχει την περιουσία των χριστιανικών ιδρυμάτων. Το 2010 σκοτώθηκαν τρει χριστιανοί στη Μαλάια, αλλά δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα η ε, υπόθεση αυτή παρά το γεγονό ότι οι πέντε δράστες είναι γνωστοί. αντιμετωπίζει τους Κούρδους σε συριακό επίπεδο. Η Τουρκία παραβιάζει την κυριαρχικότητα της Συρίας και οι χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης εκπαιδεύουν τους πεσμεργά για να αγωνιστούν εναντίον του Ισλαμικού κράτους και ήδη αυτοί οι Κούρδοι βομβαρδίζονται από την Τουρκία και σκοτώνονται. Και παρόλα αυτά εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Μα μπορεί μια τέτοια χώρα θα μπορούσε κάποτε να αποτελέσει εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που έχουμε ήδη ανακαλύψει ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει το Ισλαμικό κράτος με παραδόσεις όπλων από την Τουρκία και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι το απεκάλυψαν αυτό βρίσκονται τώρα ενώπιον του δικαστηρίου για την αποκάλυψη αυτή. Με ποιο τρόπο μπορείτε σοβαρά να πείτε ότι αυτή η χώρα μπορεί να αποτελέσει εταίρωμα, ε, εταίρος μας. Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη, καταλάβετε το. Ένα λεπτό, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα ικανοποιημένο για μια τόσο δύσκολη ε, έκθεση και για μια τόσο προβληματική χώρα αλλά ως πρόεδρος της Μικρής επιτροπής ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία πύρη τους εισηγητές των κομμάτων την κυρία ζόμερ για την πραγματικά επαγγελματική δουλειά την οποία έκαναν μέσα στις αρχές και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίσθημα ευθύνη. Βεβαίω στην έκθεση αναφέρονται πολλά από τα ελλείμματα πολιτικής που έχει η Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών χωρών να επικυρώσει το δίκαιο της του 1982 που είναι η μόνη που ένταξη χώρα που δεν το είχε επικυρώσει, να άρει την απειλή πολέμου για την Ελλάδα, να σταματήσει τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των χωρικών υδάτων των γειτονικών χωρών, να αναγνωρίσει την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και τη λειτουργία της Χάλκης, να αλλάξει την τραγική πολιτική της με πολλά θύματα στην νοτιοανατολική Τουρκία και βεβαίως δεν θα ανοίξουν τα κεφάλαια αν δεν επιβεβαιώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Merci. λεπτό πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την περιεκτική και πολύ καλά οργανωμένη έκθεση. Θα τονίσω όμως κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία που ε, κατά τη γνώμη μου είναι τα πιο σημαντικά. Σήμερα νομίζω ότι προχωράμε σε σχέση με το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο δυστυχώς έχει οδηγήσει στην ε, μείωση των μεταρρυθμίσεων και στην πρόοδο, την ε, πάυση της πρόοδου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδείνωση στην ελευθερία και ελευθερία λόγου και έκφραση στη χώρα έχει παρατηρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό και τον, ε, ε, παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει ώστε η Τουρκία να λύσει τα διμερεί θέματα με τους γειτονές της και η επιτυχία των διαπραγματεύσεων για την Κύπρο είναι πολύ σημαντική για την Ένωση αλλά και για Δεύτερον, δεν υπάρχει χρόνος να να αρνούμαθα την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Ωστόσο, έχω ανησυχίες όσον αφορά την τελευταία συμφωνία Ένωσης Τουρκίας. Ωστόσο θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την υποστήριξή μου σε όλους τους ε, Τούρκους και τις αρχές που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας και ορισμένους από τους συναδέλφους θα ήθελα να τους θυμίσω τη σοφία του λαού μου ότι ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τη δύναμη για να κρύψουμε τις προθέσεις μας. Ο εισηγητής ε, επισημαίνει δικαιολογημένα στην παράγραφο 13 της ε, βίες ε, πράξης των ε, λεόντων του Αλάχ και υπάρχει μία σχέση της ομάδας αυτής η οποία παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ανατολική Τουρκία. Ε, και νομίζω θα πρέπει να αναλυθεί δράση. Από έγκυρες πηγές ε, μου είπαν ότι η ομάδα αυτή, οι λέοντες του Ισλάμ, ε, πρέπει να προστατεύσουν τον πρόεδρο Ερντογκάν τόσο από το ΠΚΚ όσο και από άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης αυτής της ομάδας και υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για πρόσφυγες οι οποίοι είναι, από τη Συρία που είναι ιδιαίτερως εκτεθειμένοι ε, σε βασανιστήρια από αυτές τις ομάδες ενώ πίστευαν ότι επιτέλους θα είναι ασφαλείς ε, στην Τουρκία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και, Ενωμένης, ε, και Ευρώπης σε αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Σχάκη, η συμφωνία μεταξύ ε, Ένωσης και Τουρκίας ε, σηματοδοτεί ένα νέο είδος ε, δικαίου. Ειλικρινά όλες οι ανησυχίες αποτελούν πλέον ένα προβλέψιμο σχέδιο, ένα προβλέψιμο σχήμα, το οποίο όμως εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό. Και φαίνεται ότι εδώ είμαστε ο μόνος θεσμός, η μόνη πολιτική, οι μόνοι άνθρωποι που ειλικρινά και κριτά μιλάμε για το τι συμβαίνει πραγματικά. Υπό το φως των τεραστίων προβλημάτων που σωρεύονται, ακόμα πιο προβληματικό είναι ότι η Κομισιόν έχει σταματήσει στην ατζέντα της με την τελευταία έκδοση της ετήσιας της έκθεση. Συγγνώμη κυρία Σχάκε, αλλά φαίνεται να μην υπάρχει διερμηνία στα αγγλικά. Μα μιλάει στα αγγλικά η κυρία Σχάκε. Τα λέω αγγλικά, <laughs> αν για όποιους δεν κατάλαβαν. Ε, συγγνώμη, εγώ άκουσα αυτό που μου είπαν μόνο. Αλλά φυσιολογικό να μην ακούτε αγγλικά. Υπήρχε πρόβλημα διερμηνίας? Όχι, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψα, λέει η Πρόεδρος. Συνεχίζω ή τα ξαναλέω από την αρχή. Ναι, λοιπόν, ε, ας ξαναρχίσετε. Στα αγγλικά τα λέω. Λοιπόν, Πρόεδρε, συνάδελφοι, <laughs> Υπουργέ, Επίτροπε η ψήφος μας για την ετήσια έκθεση για την Τουρκία φτάνει σε ακόμα πιο χαμηλό σημείο. Το κείμενο που θέλουμε να ψηφίσουμε είναι ακόμα πιο επικριτικό όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη βία ε, νοτιοανατολικά και ειλικρινά πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο είναι προβλέψιμο αλλά όχι λιγότερο ανησυχητικό. Και μόνο η πολιτική σε, και το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης που ξεκάθαρα τα λέει όλα αυτά είμαστε εμείς. Είναι πολύ προβληματικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν σταματήσει τις ατζέντε τους. Η Κομισιόν καθυστέρησε τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης και υπήρχε μια οικοφαντική σιγή όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία πρόσφατα. Είδαμε τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν να βιάζεται να σφίξει το χέρι του Προέδρου Ερντογάν 8 μέρε πριν από κρίσιμε εκλογέ. Και μάλιστα θα ήθελα εγώ να τον δω να συμμετέχει στη συζήτηση για την Τουρκία εδώ. Ε, είναι πολύ σημαντικό που το Συμβούλιο δεν αναθέτει, να μην αναθέσει σε άλλους τις ευθύνες του για το άσυλο και να ε, ενώ θεωρεί ότι η Τουρκία θα λύσει τα προβλήματα ε, και πιστεύω ότι η συμφωνία με την Τουρκία είναι τοξική και πληρώνουμε τεράστιο τίμημα εις βάρος των αρχών μας και του λόγου μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει και ελπίζουμε ότι η Συμβούλιο και η Επιτροπή θα αλλάξουν πορεία. Ναι, καλά τα αγγλικά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει η κυρία Σχάκη. Κυρία Σακοράφα, ένα λεπτό κύριοι συνάδελφοι η έκθεση προόδου αποτυπώνει για πρώτη φορά με τόσο αποκαλυπτικό ρεαλισμό την πραγματικότητα στην τουρκία και αυτό το πιστώνεται η κυρία πύρη και όσοι συμμετείχαμε στη διαδικασία. υπογραμμίζω δύο σημεία καλείται την τουρκία να διαπραγματευτεί για συνολική και βιώσιμη λύση στο κουρδικό. όσο όμως η ευρωπαϊκή ένωση χαρακτηρίζει το πκκ τρομοκρατική οργάνωση ενώ αποτελεί μέρος τη λύση, νομιμοποιεί τι εκαθαριστικές επιχειρήσεις της τουρκίας ακόμα και μέσα στη συρία χαιρετίζετε την κοινή συμφωνία για το προσφυγικό και την εμπλοκή του νατο στο αιγαίο και πάλι η ευρωπαϊκή ένωση σκόπιμα εμπλέκει τρίτους σε ζητήματα που την αφορούν επικαλούμενη αδυναμία. η αμέσως προηγούμενη αφορά στην εμπλοκή του δουνουτού. τα αποτελέσματα θα είναι το ίδιο καταστροφικά για τους λαούς. όπου εμπλέκεται το νατο οξύνει τις εντάσεις. κλείνω με ένα ερώτημα. ποια ενταξιακή διαδικασία μπορεί να υπάρξει με μια χώρα όπως την περιγράφει η έκθεση η οποία επιπροσθέτως καταπατά το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που υπογράφει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μαραγκάλ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς υποστηρίζουμε την εκθέση τη κυρία Πύρη, η οποία έχει κριτικό χαρακτήρα όπως και θα πρέπει και υποστηρίζουμε και την ε, το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 για δύο λόγους. Η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Η Ευρώπη είναι ελλειπής χωρίς την ε, Τουρκία παρά τους τείχους που ορθώνονται και παρά την αντιδημοκρατική στάση των τωρινών τουρκικών αρχών. Είναι όμως δεδομένο ότι η διαδικασία της ένταξης έχει επιμολυνθεί με το θέμα των προσφύγων. Η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτό το θέμα ως αντίτιμο για να επιτύχει πολιτικές παραχωρήσεις. Γι' αυτό είναι αδύνατον να συζητήσει το Κοινοβούλιο για μια τέτοια συμφωνία που δεν μπορεί ούτε να την επικυρώσει ούτε να την απορρίψει. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το να απελάβουν στη Συρία η Τουρκία πολίτες που έχουν έρθει από εκεί για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε επίσης να επικροτήσουμε τη στάση της Τουρκίας εν των Κούρδων. Και οι Κούρδοι πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, αλλά πρέπει να αρθεί η κατάσταση πολιορκίας η οποία είχε σταματήσει στο παρελθόν. Δέχεστε μια μπλε κάρτα κύριε Μαραγάλ από τον κύριο Φουντούλη. Ο κύριος Συναδινός, συγγνώμη θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο γιατί θα μας κάνει εδώ να ξεχάσουμε και τη γεωγραφία πώς αποδεικνύεται ότι η τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. ευχαριστώ. Ναι, κύριε συνάδελφε, μπορείτε να κοιτάξετε την ιστορία του παρελθόντος, να δείτε το χάρτη της Ευρώπης και θα καταλάβετε ότι έχω δίκιο. Η Τουρκία είναι Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί και πρέπει να γίνει κομμάτι της Ευρώπη και η ιστορία μας δίνει πολλά παραδείγματα και πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτής της πραγματικότητας. Και η γεωγραφία ακόμα περισσότερο και η γεωστατική ακόμα περισσότερο η Ευρώπη και η Τουρκία πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση της Συρίας αυτό είναι και ένας λόγος να την αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της επίσημης Τουρκίας και της πραγματικής Τουρκίας. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Βίνμπερκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για την Τουρκία μας ε, αναφέρει πολλά γεγονότα τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσει να προβληματιστούμε λιγάκι για την κατεύθυνση που έχει πάρει αυτή η χώρα και για το αν είναι ορθό να είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι έχει σταματήσει η θετική πορεία της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες, την ελευθερία έκφρασης, συναθρίζεστε, τη λειτουργία της δημοκρατίας, έχουν χαθεί όλα αυτά. Βλέπουμε επίσης ότι παραμένει το 10% ως φράγμα στην ε, εκπροσώπηση των πολιτών στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Στα θέματα ασφάλειας, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως παιχνίδι οθωμανικών αυτοκρατορικών επιδιώξεων με ενσωμάτωση βυζαντινικού χαρακτήρα στη δράση της. Μήπως η Τουρκία όμως τελικά παίζει το παιχνίδι του Ισλαμικού κράτους. Άκουσα ή έκουσα. Μήπως έχει νόημα να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες, όπως έχουμε πράξει. Ο κύριος Τεχράφ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε, σένταξε πάλι μια πραγματικά περιττή έκθεση, μια έκθεση για τα σκουπίδια για την Τουρκία η Τουρκία πραγματικά έστειλε έστειλε πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κέρδισε πολλά χρήματα από αυτό ταυτόχρονα διεξάγεται μια, μια γενοκτονία έναντι του κορδικού λαού και η Τουρκία ε, υποστηρίζει τους Ισλαμιστές. Υπάρχει μια Ισλαμική Οθωμανική δικτατορία η οποία φροντίζει από την Κωνσταντινούπολη για τον εξισλαμισμό της χώρας κηρύττοντας το μίσος κατά της Δύσης και ε, ε, οθώντας τους πρόσφυγες να πλημμυρίσουν τα χωριά και τις πόλεις μας. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρξει χορήγηση θεώρηση ε, στην ε, Τουρκία. Η Τουρκία θα πρέπει ποτέ να μπει στην Ευρώπη. Ο κύριος Φουντούλη για ένα λεπτό. Η ονομασία έκθεση προόδου για την Τουρκία είναι ατυχή και δείχνει πω οι Ευρωπαίοι πολιτικοί εξοραίζουν την πραγματικότητα και επιθυμούν να εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα. Σε κανένα τομέα δεν έχει σημειώσει πρόοδο η Τουρκία. Αντιθέτως παραμένει πάντα ένα κράτος αλαζονικό, μακριά από κάθε έννοια σεβασμού προς τους γείτονές του, με πλήρη αδιαφορία προς το διεθνές δίκαιο. γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως η τουρκική κυβέρνηση υποστήριξε τους εγκληματίες του ισλαμικού χαλιφάτου που συνεχίζει εδώ και 42 χρόνια να κατέχει παράνομα τμήμα της κύπρου και κάθε μέρα προβάλλει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον της ελλάδος. στο θέμα του μεταναστευτικού την ίδια μέρα που επαναπροωθήθηκαν 150 μετανάστες προς την τουρκία έφτασαν στα ελληνικά νησιά 600. η τουρκία κάνει τα στραβά μάτια ή συνεργάζεται με τους δουλέμπορους και μία από αυτέ τι ενέργειε θα αρκούσε για να έχει διακοπεί προπολού κάθε σκέψη για συνεργασία με αυτό το κράτο. Αντιθέτω όμω η ένωση επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο την τουρκία με ένα καθεστώ που φυλακίζει όποιο τολμά να το αμφισβητήσει. τελευταία μάλιστα αποφάσισε να σέρνει στα δικαστήρια και δημοσιογράφου άλλων χωρών αν τολμούν να σατυρίζουν τον μεγάλο σουλτάνο ερντογάν με τη συμπαράσταση βεβαίω και τη καγκελαρίου μέρκελ που μάλλον σκέφτηκε πω είναι πολλοί οι τούρκοι ψηφοφόροι στη γερμανία. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ στηρίζω την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε το ρόλο της Τουρκίας στην υποδοχή με αξιοπρέπεια τριών εκατομμυρίων προσφύγων. Θα πρέπει ωστόσο να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για την ελευθερία έκφραση στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου καθώς και για την ανθρωπιστική κατάσταση και την δυσανάλογη στρατητική αντίδραση στην ανατολική πλευρά τη χώρα. Θα πρέπει και οι δύο πλευρέ να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Επίση, καλωσορίζω το πρόγραμμα δράση τη Ένωση με την Τουρκία και την απελευθέρωση 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά όλα θα πρέπει να εφαλίσουν του πρόσφυγε. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τι διεθνεί προδιαγραφέ και την αρχή τη μία απόθεση. Non refoulement. Η Τουρκία θα πρέπει να καταγραφεί ως ασφαλής χώρα επιστροφής. καλύτερο τρόπο για να προωθηθούν οι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει είναι ανοίγοντα κεφάλαια με, για ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν είναι παζάρι, κυρία Πρόεδρε, είναι win-win κατάσταση. Χαουίτε, ένα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, η έκθεση αυτή ηθελημένα δεν κρίνει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για του πρόσφυγε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η συμφωνία αυτή έχει θεωρηθεί παράνομη και μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι σωστό η Ευρώπη να προσπαθεί να συνεργαστεί με την Τουρκία και με όλες τις χώρες που γειτονεύουμε τη Συρία στην ανθρωπιστική προσπάθεια για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Μόνο όμως όταν αυτό σημαίνει πλήρη σεβασμό για το διεθνή, ε, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει ε, την δημοκρατία. Εγώ πήγα πριν από ένα μήνα στην Νότια Ανατολική Τουρκία ε, ε, μπορείς να πολεμάς τους τρομοκράτες αλλά όχι τους δικούς σου, το λαό σου να επιτρέπεις ε, να ταφούν οι άνθρωποι και να επιστρέφονται σε μέσα σε μια διαδικασία ειρήνευσης με τους Κούρδους και μην ε, χώνεις τη στενή τους φίλους, τους δημοσιογράφους επειδή μιλούν, λένε τα όσα συμβαίνουν δεν θα έπρεπε να έχεις τίποτα να κρύψεις το Υπουργείο Δικαιοσύνη λέει πω αυτοί που κατηγορούνται για τρομοκρατία θα του αρθεί η εθνικότητα. Αυτό είναι. σημαίνει ότι αψηφάς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το συγκεκριμένο το άρθρο 15 της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να καταλάβεις ε, πόσο μειοπικά είναι όλα αυτά τα επιχειρήματα και αν η Τουρκία υποκρίνεται θα πρέπει και εμείς να υποκριθούμε. Ευχαριστώ κύριος Μπασίρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν ο οποίος βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις και ζητά κάποιον να του δώσει βοήθεια, αλλά αυτός που θέλει να τον βοηθήσει ζητά ένα αντίτυπο. Αυτό συμβαίνει και με την Τουρκία. Και φαίνεται ότι πολλοί συνάδελφοι εκπλήσονται από αυτό το γεγονός. Ιδανικά και εγώ θα προτιμούσα να είχαμε διαχωρίσει όλα αυτά τα θέματα μεταξύ τους, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Η Τουρκία διαδραματίζει γεωπολιτικά ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή και χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους <clears throat> για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συστηματικά θέματα τα οποία είναι μεγάλη σημασία για όλους μας από το πακέτο μετανάστευσης μέχρι και τη συνομιλία ένταξης. Όλα τα θέματα αυτά δίρυτα επικαλύπτονται αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας τρομοκρατεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μεν και να μην δώσουμε απόλυτη ελευθερία στην Τουρκία, αλλά <clears throat> συγχρόνως πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι χρήσιμη και απαραίτητη για μας για θέματα όπως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε την σχέση μας και όχι ένα βήμα προς τα πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την έκθεση του 2015 για την Τουρκία μπορούμε να υπογραμμίσουμε με σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η συνεργασία στο προσφυγικό και τα θέματα της ε, ειρήνευσης στην Κύπρο. Είναι απαραίτητο να ενοιχτούν τα νέα κεφάλαια όταν εκπληρωθούν οι προδιαγραφές, τα benchmarks και επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε θεματικά ζητήματα η κατάσταση ασφάλισης στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί το 2015 για τα οικονομικά ε, θέματα χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες. Λόγω της τωρινής γεωπολιτικής κατάστασης πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία των δύο πλευρών για τη μετανάστευση. Παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της μετανάστευσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις κοινέ δράσεις με πραγματιστικό τρόπο προς αμοιβαίο, αμοιβαίο όφελος. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει στις συνομιλίε για την επανένωση της ε, Κύπρου που θα οδηγήσει σε ωφέλη και στις δύο κοινότητες. Γενικά μπορούμε να δούμε ότι η διαδικασία της Τουρκίας προχωρά. Ρίτ για ένα λεπτό. Ε, πρόεδρε, η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική αυτή καθ' αυτή και ιδιαίτερα τώρα εν ώψη του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό, επιτρέπει στον Ερντογκάν να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Η Τουρκία δεν είναι τμήμα της Ευρώπης. Ε, το 98% της χώρας βρίσκεται στην Ασία. Και ενώ η Ευρώπη έχει μία η Τουρκία δεν είναι τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ε, η ναι μεν η Τουρκία έχει γίνει ένα κοσμικό λαϊκό κράτος αλλά αυξάνονται όλο και περισσότερο οι τάσεις εξισλαμισμού. Τι θα σημαίνει αν προσχωρήσει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, ακόμα και τα δεδομένα για τον πληθυσμό δεν είναι ακριβή. Μέχρι 79 εκατομμύρια φτάνουν και όταν η Τουρκία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι πρόσφυγες, τα 2,5 εκατομμύρια θα έχουν το δικαίωμα να μεταβούν στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Τόρις είναι μέλη των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστικών, ένα πανευρωπαϊκό ε, κόμμα ε, στο οποίο συμμετέχει. Ε, η συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από χρόνο λόγος για την Μεγάλη Βρετανία να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο κύριος Σαφχάουζερ για ένα λεπτό. Ε, πρόκειται για μια εξαιρετικά διαυγή, έκθεση η οποία αποκαλύπτει αλήθειες για τον δικτάτορα Αρντογκάν. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα μάτια μπροστά σε κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να αναμένουμε ε, την άμεση πάυση των συμφωνιών του Όσλο. Όχι, η έκθεση αυτή προτείνει την επανεκκίνηση αυτού του διαλόγου. Κυρίε και κύριοι, θέλετε ένα πολιτικό Ισλάμ στην Ευρώπη, τον προπικανδισμό του Ισλάμ, γιατί φοβούμε ότι πράγματι αντιμετωπίζεται την αλήθεια ενό ε, τρομοκρατικού, ενός, ε, μιας χώρας που ενισχύει τον ίσις ένα μαφιώσικο καθεστώς ε, το οποίο ε, παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ ώψη αυτής της αλήθειας, της πραγματικότητας επιλέξατε το ψέμα ε, απέναντι σε έναν εκβιαστή ψεύτη ο οποίος τελικά εκβιάζει τους λαούς. Ε, ε, Η Τουρκία είναι και θα είναι ε, γειτονάς μας και ε, βεβαίω ασφαλώ θα έπρεπε να αναζητήσουμε σχέσει καλή γειτονία. Ωστόσο, ένα καλό γείτονα σέβεται τι μέσει που έχει αναλάβει, τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση και δεν αντιδρά με επιθετικότητα στην άσκηση κριτική. Ε, αναμένω να σεβαστείτε τι ε, συμφωνίε ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ανοίξετε νέε μεταναστευτικού οδού. Η το ευρωπαϊκό τμήμα της ε, Τουρκίας περνάει από την ε, αναγνώριση της ε, τουρκικής ηθαγένειας των ε, πολιτών στην ε, Βουλγαρία, στο Παύλοβο. Η τήρηση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων σημαίνει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Βουλγαρία, πρόσβαση στα μέσα μαζική ενημέρωση τη Βουλγαρία και δικαίωμα αυτοδιάθεση. Η Τουρκία επίση ε, προσπαθεί να επηρεάσει τι εξελίξει στο Αζερβαϊτζάν. как Πώς ε, θα σχολιάζατε την ε, τήρηση της συμφωνίας δεδομένου ότι η Βουλγαρία συνέλαβε 97 παράνομους μετανάστες χθες. Δεύτερον, πώς ε, θα σχολιάζετε την απαράδεκτη παρέμβαση της Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Βουλγαρίας ε, ενορχιστρώνοντας κάποιες πολιτικές διαδικασίες εντός της χώρας αυτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι γείτονες θα έπρεπε πάντοτε να έχουν τα, τις ε, μυστικές τους πληροφορίες και τα εργαλεία για να μπορούν να επηρεάζουν τις γειτονικές χώρες και πρόκειται για την ευθύνη αυτών των ειδικών υπηρεσιών, δηλαδή προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να αναχαιτήσουν τέτοιου είδου προσπάθειε, είτε πρόκειται από την Τουρκία, είτε από τη Ρωσία, είτε από οπουδήποτε αλλού. Όσον αφορά τη συμφωνία αυτή, θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι αναμένω ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει το άνοιγμα μια νέα μεταναστευτική διόδου μέσω των Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κάτι Πύρη γιατί η αποτύπωση της κατάστασης που μας έδωσε στην έκθεση είναι απολύτως ακριβής. Για μα η ετήσια αυτή έκθεση δεν είναι μια ευκαιρία να κατηγορήσουμε την Τουρκία. Και η επισήμανση ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, δικαιοσύνης και θρησκευτικών ελευθεριών λαμβάνει το πραγματικό της νόημα μόνο αν αποτελέσει το έναυσμα για μια βαθιά συζήτηση και με την τουρκική κυβέρνηση αλλά και με την κοινωνία των πολιτών η οποία διστακτικά πια συνεχίζει να έχει σαν όραμά της την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όμως είναι, επιτέλους πρέπει να προχωρήσει μια πολιτική λύση στο κουρδικό με μονομερή κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονη λήξη των αστυνομικών επιχειρήσεων πριν ε, πράξεις όπως η άρση της βουλευτική ασυλίας που προωθεί η κυβέρνηση οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες μέρες. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαρνέσκι για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ας κλείσουμε τα μάτια μας. Ας φανταστούμε το χάρτη της Ευρώπης μετά από την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γειτονές μας ήταν το Ιράκ, το Ιράν και η Συρία. Δεν είναι συναρπαστική αυτή η γειτονιά. Κυρίε και κύριοι, ελπίζω ότι στη συζήτησή μας θα αποφύγουμε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά οι ίδιοι πολιτικοί που όλα αυτά τα χρόνια θεωρούν ότι εμείς δεν θα πρέπει να δεχτούμε την Τουρκία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτοί οι ίδιοι πολιτικοί έχουν υπογράψει μια συμφωνία με την Τουρκία για την επανεισδοχή προσφύγων. Αυτό γιατί υπήρχε μια πολιτική ανάγκη με τις τοπικές εκλογές σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να μιλάμε με τον τρόπο αυτό για την Τουρκία υπό το φως των τοπικών εκλογών. Δέχεστε μια μπλε κάρτα κύριε Ελτσέτ. Κύριε Κάρβερ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Τσανέσκι. Κανείς δεν μιλάει για το γεγονός ότι έχει αλλάξει και η αντιμετώπιση σε αυτό το κοινοβούλιο. Αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πληθυσμό 77 εκατομμυρίων περίπου θα έχει το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών και οι τωρινέ χώρε μέλη θα έχουν ακόμα λιγότερου βουλευτέ. Μήπω είναι και αυτό ένα λόγο να κρατήσουμε την Τουρκία εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όλες οι χώρες μας θα έχουν ακόμα μικρότερη δημοκρατική εκπροσώπηση. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο δεξέχων βουλευτής ο οποίος έλαβε το λόγο θεωρεί ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επεκταθεί παρά μόνο με το να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Δεν σημαίνει τίποτα τέτοιο. Μπορούμε να έχουμε κάποια προσαρμογή και κάποια σχετική μείωση των μελών από τα τωρινά κράτη-μέλη ακολουθώντας τους κανόνες που λένε ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε σε 751 βουλευτές. Η κυρία Φωνστόρκ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε σήμερα για το νέο καλό φίλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Μετά από τη συμφωνία για τους πρόσφυγες θα ακολουθήσει η ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς βίζα και μετά η προσχώρηση. Μα δεν υπάρχει κανένα στην Ευρώπη που βλέπει την κατάσταση στην Τουρκία για τα δικαιώματα συναθρίζεστε, ε, ελευθερία του τύπου, τα δικαιώματα των γυναικών, όλα αυτά καταπατώνται από τον πρόεδρο Ερντογάν και με τα δύο πόδια του. Όλοι οι αναλυτές έχουν απόλυτη ομόνια ότι εμείς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάτι καλό με την προσέγγιση αυτή προς την Τουρκία. Νομίζετε ότι θα κάνει τη βρώμικη δουλειά για μας η Τουρκία για να κρατήσει η κυρία Μέρκελ τα ανοιχτά τη σύνορα. Η Τουρκία είναι μια χώρα χωρίς ε, ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς ελευθερία του συναθρίζεστε, χωρίς ελευθερία του τύπου. Τα δικαιώματα των χριστιανών, των μειονοτήτων, των Κούρδων παραβιάζονται κάθε μέρα ή αντιμετωπίζονται με βία από την αστυνομία. Ο Ερντογάν έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά του δικού του πληθυσμού και επίσης εναντίον των γειτονικών χωρών. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να είναι ουσιαστικά η απόλυτη ομολογία αδυναμίας της Ευρώπης να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να επαφίεται σε μια χώρα σαν την Τουρκία. Αυτό είναι πραγματικά παράλογο. Η Τουρκία δεν δέχεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Όπως είπε ο κ. Σέντογαν, η δημοκρατία είναι ένα τρένο από το οποίο μπορούμε να βγούμε. Οι ε, μιναρέδες είναι οι, οι λόγχες μας και τα τζαμιά είναι οι στρατώνες μας. Δεν μπορούμε, αυτά λέει ο κ. Σεντογάν, δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε απλώς διακοπή των σχέσεων με την Τουρκία. Πρέπει να τη σταματήσουμε μια και για πάντα και να μην υπάρξει ποτέ προσχώρηση αυτής της χώρας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Φωνστόκλε, Πρόεδρος. Ωραία τα λέτε για τον κύριο Ερντογάν και είναι ενδιαφέρον να σας δει κανείς σε αυτήν την πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Ο επόμενος ομιλητής ο κ. Μπρός για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Επειδή η Τουρκία χρησιμοποιεί το πετρέλαιο που βγαίνει από τα, ισλαμικά, από τα δηληστήρια του Ισλαμικού κράτους επειδή έχει δώσει υλικό που απαραίτητο για την επεξεργασία του αερίου Σαρίν επειδή βομβαρδίζει τους αντάρτες Κούρδους αντί να βομβαρδίζει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους επειδή η Τουρκία αφήνει τους ε, μετανάστες που είναι στο έδαφος να μπαίνουν παράνομα στο χώρο Σέγγιν. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαράδεκτο να απελευθερωθούν οι θεωρήσεις Τούρκων πολιτών που έρχονται στην Ευρώπη, καθώς είναι απαράδεκτο επίσης να δοθούν τρία δις επιπλέον στην Τουρκία και πάνω απ' όλα θα ήταν πραγματικά αυτοκτονικό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Εκτιμώ ε, βέβαια ότι η Τουρκία είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Εκτιμώ τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας για να, λύσουν, ε, να λύσει το προσφυγικό και ακριβώ τώρα με αυτή τη συνεργασία θέλω να διαμαρτυρηθώ κατά της βίας που ασκεί η Τουρκία κατά των Τούρκων. Αυτό γίνεται και στην επικράτεια της Τουρκίας. Σας θυμηθούμε ότι βομβαρδίζει τα κουρδικά στρατόπεδα στο Ιράκ, στο Κόμπανι στη Συρία, η κλιμάκωση της ε, κατάστασης ε, τονίζεται από την αντίδραση του ΠΚΚ ε, που αντιδρά στην τρομοκρατία του κρατικού κράτους. Η Τουρκία έχει πάψει να λέει τους Κούρδους, να αποκαλεί τους Κούρδους Τούρκους του βουνού. Το τουρκικό κοινό ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για την τραγική ιστορία του, τουρκικού εθνικισμού όπως ε, την γενοκτονία που θα ε, εορταστεί την επόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ πολύ. Η ρύθμιση τη σχέση με την Τουρκία είναι ένα από τα σημαντικότερα μελήματα τη ε, Ευρωπαϊκή Κομισιόν, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερω κρίσιμη και βεβαίω εγκαιμονεί πάρα πολλού κινδύνου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι ανησυχητικά, όπως για παράδειγμα το κουρδικό. Η παρούσα κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί με την ε, βία να επιλύσει το θέμα αυτό και μάλιστα να πάρει ε, λευκή κάρτα για να το κάνει. Οι συνθήκε που αποκρατούν είναι συνθήκε εμφυλίου στην Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμφωνο με εμά, δεν μπορεί να μα βρει σύμφωνο. Η έκθεση στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να προσπαθήσει να διαδραματίσει το ρόλο ενός διαμεσολαβητή. Το πρότυπο θα μπορούσε να είναι η ειρηνευτική Συμφωνία στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου όλα τα ενεχόμενα μέρη κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακόμα και εκείνα που τα θεωρούσαν τότε ή τα είχαν κατατάξει στους τρομοκράτες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Θεοχάρους για ένα λεπτό τόσο η έκθεση όσο και πλήστοι συνάδελφοι λένε ξεκάθαρα ότι η τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης παρά τις δήθεν θετικές εξελίξεις στο κυπριακό όπου βέβαια πρόκειται για πλάνη επίτροπε χαν και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα διαπράξει μέγα λάθος αν γίνει συνεργός σε διαδικασίες που προάγουν την τουρκική επιθετικότητα εναντίον της κυπριακής δημοκρατίας και ανατρέπουν αποφάσεις του ιδίου της επιτροπής και του συμβουλίου αν πιστεύετε ότι επίκειται λύση δηλώνω ότι λύση αυτή τη στιγμή, τη στιγμή σημαίνει διάλυση της κυπριακής δημοκρατίας διότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και η αρχή της και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όρια σύμβατη. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αντί να υπερασπίζεται την κυπριακή δημοκρατία απορρίπτει τροπολογίες που την στηρίζουν στη λογική της επικείμενης λύσης και της εκλειπούσας κυπριακής δημοκρατίας. Ακόμη και η Επίτροπος δεν χρησιμοποιούσε, η Υπουργός ούτε μια φορά δεν χρησιμοποίησε τον όρο Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ευθύνη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ο τρόπος και η μορφή της λύσης του κυπριακού είναι όμως καθήκον του να διαφυλάξει ως θεματοφύλακας των αρχών και αξιών της ευρωπαϊκής ένωσης και να διασφαλίσει ότι η λύση θα σέβεται τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς παρεκκλήσεις για όλους τους πολίτες. εν εναντία περιπτώσει θα είναι συνυπεύθυνο για την απόρριψη της λύσης από τον κυπριακό λαό. γι' αυτό σας καλώ να απορρίψετε την έκθεση. ευχαριστώ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 Ε, και δείχνει το πώς αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη. Αλλά αυτό έθεσε και τους ε, Τούρκους κάτω από πίεση. Η Άγγελα Μέρκελ χρησιμοποίησε τη φράση «Είμαι Σαρλί» και δείχνει πως ε, εμείς οι ευρωπαϊκοί ηγέτες αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ε, θέματα και είμαστε ε, στο έλεος των εκβιασμών. Μάλλον θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας παρά να παραμείνουμε εξαρτημένοι από κάποιον όπως είναι ο Ορντογάν. Eh, Κυρία Λάγκε, ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, η συγκίτρια βρίσκεται σε μια πολύ δυσχερή θέση το προηγούμενο χρόνο, στην προηγούμενη έκθεση υπήρχαν διάφορες ε, φράσεις οι οποίες στη τελευταία στιγμή αφαιρέθηκαν που αφορούσαν το άνοιγμα διαφόρων κεφαλαίων και τις διαπραγματεύσεις. Εδώ δεν, ε, τώρα πια δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεκινήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, υπάρχουν, περιστέλλονται πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά στην έκθεση αυτή Παρόλα αυτά επισημαίνουμε και πάλι στις ε, τις διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει, έχει αλλάξει όμως γύρω μας ε, ο κόσμος. Πολλοί συνάδελφοι το επισημαίνουν. Δεν θα πρέπει να συνδέσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με τις διαπραγματεύσεις ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, η δική μου ομάδα θα στην την έκθεση γιατί δεν επιθυμούμε το άνοιγμα περαιτέρω ε, κεφαλαίων. Ε, ο, προ, ο πρόεδρος Τουρκίας δεν επιθυμεί να τον σατυρίζουν και βλέπουμε ποια απόσταση το χωρίζει από την Ευρώπη. Η κυρία Καηλία έχει το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι και επίτροπε λόγω της προσφυγικής κρίσης συνδιαλεγόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο με την τουρκία αν και δεν φαίνεται η συμφωνία να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι δεν δώσαμε λευκή επιταγή και πως απαιτείται σεβασμός στις ζωές των προσφύγων αλλά και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει η τουρκία να σέβεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την ανεξαρτησία των αρχών αλλά και τα μειωνοτικά δικαιώματα των κούρδων να σέβεται την εθνική κυριαρχία των γειτόνων της καθώς παρατηρούμε καθημερινά προκλητικές παραβιάσεις στο αιγαίο επιτέλους να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα από την κύπρο και φυσικά αναμένουμε την αναγνώριση ιστορικών γεγονότων της γενοκτονίας των ποντίων των αρμενίων και των ασσυρίων. επιπλέον πρέπει η τουρκία να σέβεται τις ιστορικές μας εκκλησίες Λειτουργώντα τεσός μουσεία και όχι ως τζαμιά όπως στην Αγία Σοφία Τραπεζούντας και πολλά άλλα. Η Τουρκία έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τη. Πρέπει να προχωρήσει σε πάρα πολλέ μεταρρυθμίσει για να χτιστεί και πάλι η εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κρίστα Μπάτεφ, Εθνικό Ήρωας και ιδιοφυΐα της Βουλγαρίας ε, ρώτησε, ε, με αποκάλεσε την, Ευρώπη, την Τουρκία την Οθωμανική τότε τον ε, ασθενή της, Ευ... της Ευρώπης. Αυτός ο άνθρωπος πυροβολήθηκε από τους Τούρκους Οθωμανούς και σκοτώθηκε και αυτή τη στιγμή η Τουρκία κρατάει στο χέρι της ολόκληρη την Ευρώπη για το αέριο, για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες. Εγώ λέω όμως ότι η Τουρκία εξαρτάται από εμά, από τα δικά μας λεφτά, από τις δικές μας αγορές και από την καλή μας βούληση. Δεν έχει άλλους φίλους, η ΙΠΑ, η Ρωσία, το Ιράν, το Ισραήλ είναι εχθροί της Τουρκίας και του Ερδογάν και είναι τώρα η σωστή στιγμή να διαλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είδους Τουρκία επιθυμεί. Η Βουλγαρία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία απελευθερώθηκε από το τουρκικό σηκώ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Τουρκίας σε ολόκληρη της την ιστορία. Η Βουλγαρία μπορεί να ηγηθεί στη μελλοντική διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μπορέσω να συνοψίσω το έργο της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων και της συζήτηση, θα έλεγα κουράγιο, α την κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, έχοντα ανοίξει 17 κεφάλαια για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1997, εσείς οι σοσιαλιστές, το ΕΛΚ, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι, θεσπίσατε μια σειρά κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχετε παραγνωρίσει ότι υπήρχε παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της, ε, υπήρχε η κατοχή της Κύπρου από το 1974 αλλά δεν έχουμε πια να δώσουμε μαθήματα στην Τουρκία γιατί η Ευρώπη και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος το οποίο περιφρονεί τους πολίτες της Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Χριστοφόρο, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σε αυτή την έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθήκο να μιλήσει ξεκάθαρα για το θέμα της Τουρκίας. Κάθε χρόνο και χειρότερα είναι η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Η ίδια η Τουρκία χειροτερεύει τη θέση τη σε όλου του θεσμού, σε όλα τα επίπεδα. Δεν σέβεται κανένα, ούτε ακόμα και τι αρχέ και τι αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση, για τι οποίε τάχατε θέλει να σεβαστεί εντασσόμενη πλήρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αν έχει κάποιο υπεύθυνο για την ενταξιακή πορεία τη Τουρκία, είναι η ίδια η Τουρκία. Θεωρώ όμω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ιδιαίτερα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι δεν μπορούν να γίνονται εκπτώσει σε αυτού οι οποίοι δεν σέβονται καμιά αρχή, ιδιαίτερα για την ενταξιακή πορεία γιατί αυτό από μόνο του θα καταργήσει την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση που είναι ένωση αρχών και αξιών και πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όσους συναδέλφους επιχειρούν και ζητούν άνοιγμα κεφαλαίου για την τουρκία πριν να εφαρμόσει τα ελάχιστα που οφείλει να εφαρμόσει. να θυμίσω ότι δεν αναγνωρίζει την ίδια την υπογραφή τη στο πρωτόκολλο τη Άγκυρα, δεν αναγνωρίζει χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει έδαφο χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρα μέλου τη Ευρωζώνη, η ίδια η τουρκία διατηρεί 40.000 στρατεύματα σε χώρα μέλος τη ευρωπαϊκής ένωσης και ήθελα να ρωτήσω τους αγαπητούς συναδέλφους τι θα έπραξαν οι ίδιοι αν βρισκόντουσαν στην ίδια μοίρα που βρίσκεται σήμερα ο κυπριακό λαός όσον αφορά τη συμπεριφορά την αντιμετώπιση και την παραβίαση αρχών από την τουρκία. γι' αυτό κύριε πρόεδρε τελειώνοντας θα καλέσω και την ευρωπαϊκή επιτροπή και τους αγαπητούς συναδέλφους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να στείλουν αυτό το ισχυρό ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπτώσεις για το θέμα της τουρκίας. Ε, ε, σας παρακαλώ όμως να τηρήσετε το χρόνο ομίλια σας και να μην το ξεπερνάτε. Ο κύριος Λόπες, θέλω να αναγνωρίσω το εξαιρετικό έργο της εισηγήτριας της κυρίας ε, Πύρη. Η Τουρκία είναι στρατηγικό εταίρο για όλε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μα κάνει να σταματούμε να μιλάμε για αυτό που είναι σήμερα η Τουρκία με την ε, ολίσθηση προς αυταρχικό κράτος του Ερδογάν με μια χώρα η οποία εν μέρη βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο με ένα κράτος δικαίου το οποίο έχει διαλυθεί με κλειστές εφημερίδες, με δημοσιογράφους στη φυλακή με τις ελευθερίες περικοπμένες για πάρα πολλούς Τούρκους και φαίνεται ότι θέλει να επεκτείνει αυτό και σε ένα χιουμορίστα γερμανό ο κύριος ε, Ερντογάν. Τι θέλουμε, να ανοίξουμε το κεφάλι 23-24 για να βοηθήσουμε τον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραβιάζονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως ανταλλακτικό νόμισμα τους πρόσφυγες για να δώσουμε ανταλλάγματα στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τι σχέσει με την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ η τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και διατηρεί το κάζους μπέλι κατά της ελλάδας. ταυτόχρονα τα τουρκικά στρατεύματα συνεχίζουν να κατέχουν παράνομα το 37% του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας. η τουρκία συνεργάζεται με τον νταές κάνει business με τους λαθρέμπορους πετρελαίου τζιχαντιστές εξοπλίζει τον νταές στη συρία και στη λιβύη. ταυτόχρονα καθοδηγεί τα δουλεμπορικά κυκλώματα που έχουν γεμίσει την ελλάδα με χιλιάδες πρόσφυγες παρ' όλα αυτά κύριε Χάν, η ευρωπαϊκή ένωση τελικά δίνει συγχωροχάρτη στην άγκυρα και την επιβραβεύει δίνοντάς της από πάνω πρίκα έξι δισεκατομμύρια ευρώ αναβαθμίζοντας την τουρκία στο πολιτικό διάλογο και καταργώντας τη βίζα για τους τούρκους πολίτες που κατά εκατομμύρια θα κατακλείσουν πλέον την ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ένωση. Κύριε Χάν, πρέπει να το καταλάβετε. Η Τουρκία δεν είναι μέρος της λύσης. Η Τουρκία είναι μέρος του προβλήματος, όπως ήταν άλλωστε και στο παρελθόν όταν διέπραξε τη γενοκτονία των ποντίων αδελφών μας γεγονός που δεν αναφέρει καν η έκθεση αν και όφιλε να το πράξει. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Παπαδάκης έχει λόγο είναι κατ' επανάληψη που επικρίνεται η τουρκία σε αυτήν την αίθουσα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών τη για φήμωση του τύπου και των μέσων κοινωνική δικτύωση για τη στάση τη στο κουρδικό για τι σχέσει τη με το Άισι, για του εκβιασμού για το προσφυγικό για την κατοχή στην κύπρο. το ερώτημα είναι ένα και πολύ απλό έχει σημειώσει πρόοδο η τουρκία όλα αυτά τα χρόνια ή πηγαίνει προ το χειρότερο; και όλοι ξέρουμε την απάντηση καθημερινά απομακρύνεται από τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης. δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα η ευρώπη να αλλάξει τη στάση χαϊδέματος της άγκυρας για να αναγκαστεί η τουρκία να γίνει μια πραγματικά δημοκρατική χώρα χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και να γίνει πόλος ειρήνης και σταθερότητας; το κολέγιο των επιτρόπων αποφάσισε χθε όπως μετονομάσει τη task force για τους τουρκοκυπρίους σε ομάδα στήριξης για τη λύση του κυπριακού. εάν πραγματικά θέλετε επίλυση του κυπριακού ένας είναι ο δρόμος αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων εφαρμογή των τεσσάρων βασικών ελευθεριών και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια σε μια ενωμένη ευρώπη. διαφορετικά οτιδήποτε άλλο θα αποτύχει. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Τζαμπάσκι έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τη εφετινή έκθεση πρόοδου για την Τουρκία είναι απαράδεκτη. Εγώ εξοργίζομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ιδέα η, τα τουρκικά να γίνει επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι απειλή προς την κυριαρχικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τη δική μου χώρα και θα έχει αποτελέσματα που δεν μπορούν να στραφούν. Εμείς υποστηρίζουμε την Ένωση της Τουρκίας, αλλά οι συνάδελφοί μας δεν το υποστηρίζουν αυτό, γιατί η Τουρκία κατέχει την Τουρκία. Θα πρέπει να παρεμβαίνουμε με τέτοιο τρόπο στα εσωτερικά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Τουρκία και κάνει την πάπια σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία της Τουρκίας στα θέματα των προσφύγων. Δεν μπορούμε να δούμε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία οργανώνει τα μεταναστευτικά ρεύματα για να μας πιέσει. Η Τουρκία επίσης <clears throat> παρεμβαίνει στα θέματα της χώρας μου και δημιουργεί πολιτικά κόμματα στη χώρα μου. Δεν λέει τίποτα το ψήφισμα για την Τουρκία που βοηθάει ξένους τρομοκράτες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λεφτά και υλικό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν να καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Η Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα καταψηφίσω. Ο κύριος Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Σωστά η έκθεση αναγνωρίζει ότι η Τουρκία είναι κέριος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η διμερή σχέση μας έχει πολύ δυνατότητα ανάπτυξης, η οποία μπορεί να πιευθεί μονάχα μέσα από μια αξιόπιστη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Φοβάμαι όμως ότι δεν συμφωνώ με την εισηγητρία σε ό,τι αφορά το τι σημαίνει αξιοπιστία για να διαπραγματευτούμε τόσο μεγάλο διάστημα με μια χώρα που δεν τη βλέπουν θετικά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι καθόλου αξιόπιστο μπορούν να κρατήσουν ακόμα δεκαετίες οι διαπραγματεύσεις στην Τουρκία και μάλλον δεν θα καταλήξουν ποτέ σε μια ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι άξιο απορίας αν μπορεί μια Ισλαμική χώρα να είναι δημοκρατική με τα ευρωπαϊκά μέτρα. Και αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιδιώξουμε Γιατί σε ευρωπαϊκές κοινωνίες χρειάστηκαν χρόνια για να οριμάσουν στο επίπεδο που είναι σήμερα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και με την καλύτερη θέληση στον κόσμο η Τουρκία θα μπορέσει σε ένα σύντομο διάστημα να καταλήξει σε μια δημοκρατική κοινωνία με τα δυτικά πρότυπα. Η διαδικασία catch the eye. Και έχει το λόγο Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο της συζήτησης αυτής κατά πολύ. Θα δώσω το λόγο μόνο σε ένα εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα. Ξεκινώ με τον κύριο Μπουσόλη. Πρόεδρε, πριν να είμαι υποψήφιος στην Ευρωπαϊκή, πριν ε, ε, πέρα από το ότι είναι ε, υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και στρατηγικός εταίρος η Τουρκία με τον οποίο πρέπει να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε τους ε, τρομοκράτες και για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του προσφυγικού και καλωσορίζω την πρόσφατη συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως θέλω να τονίσω ότι η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ένωση σχεδιάζεται στενά με την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεχάγης. Γι' αυτό η Τουρκία πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο ε, προς τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίσει τον χωρισμό των εξουσιών, τη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την ανεξιθρησκεία. Γι' αυτό θα πρέπει η Τουρκία να κάνει, βάλει σοβαρές προσπάθειες και για την επίλυση του Κυπριακού. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αρκετέ πραγματικότητε και αλήθειε για το τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία, ιδίω σε σχέση με του Κούρδου. Όμω το ερώτημα που θέτω για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια είναι το τι κάνουμε σήμερα για την Τουρκία. Θα σα πάρω κύριε Επίτροπε μερικά χρόνια πίσω. Το 2005 η Κυπριακή Δημοκρατία συνένεσε στο άνοιγμα κεφαλαίων για την Τουρκία και στι ενταξιακέ τη από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν έντεκα χρόνια. αντικειμενική διαπίστωση από όλους ανεξαιρέτως τα πράγματα στην τουρκία είναι τρεις χειρότερα από ό,τι ήταν. παραβιάσεις ελευθερία τύπου όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. σε σχέση με την κύπρο τίποτα. απαιτεί από τον ακιντζή τον τουρκοκύπριο ηγέτη να νομιμοποιήσει τους έπικους φτιάχνει φράγμα στην επαρχία της κερίνιας που είναι κατεχόμενη και από εκεί προέρχομαι εγώ ως πρόσφυγας προσπαθεί να συνδέσει με αγωγό από την τουρκία το κατεχόμενο τμήμα της κύπρου ε, αυτό σημαίνει ότι δεν επιθυμεί λύση. τελειώνω με μια υπόδειξη κύριε πρόεδρε άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την κύπρο αυτό θα σημαίνει ότι θέλει λύση. Ε, ε, ο κύριος Σεγιακό. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκή Υπήρου έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσει κάθε χώρα που θέλει να γίνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Λέσχη. Δεν πρέπει να κάνουμε παραχωρήσει και εκτόσει σε κανένα. Και αυτό ισχύει και για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι εταίρος μας, είναι στρατηγικός μας εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλά θέματα. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις για αυτό το λόγο στην Τουρκία. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας. Όλες οι χώρες που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σεβαστεί αυτές τις αξίες. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία και για τα θέματα των μεταναστών. Οποιαδήποτε χώρα φροντίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες χρειάζεται τη βοήθειά μας, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία θα πρέπει να, υποσ... να υφίσταται τις προϋποθέσεις όπως όλοι οι άλλοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σωστά καταγγέλλεται στην έκθεση παραβιάση σε μελωδό δικαιωμάτων, η διάλυση του κράτους δικαίου, και η διώξη εναντίον των κούρδων των δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών στην τουρκία. αφού όμω αναγνωρίζουμε πω η τουρκία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι βασικέ ελευθερίε ακόμα και του ίδιου του λαού τη πώ δικαιολογούνται οι πιέσει για άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24. είναι ένα σχήμα οξύμορο που φανερώνει πω κάποιοι κλείνουν τα μάτια και ενισχύουν την κρατική τρομοκρατία. έπειτα πώ ζητάτε άνοιγμα των κεφαλαίων όταν η τουρκία συνεχίζει προκλητικά να μην αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία και να καταπατά τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. είναι απαράδεκτο επίση να προωθούν τα ανταλλάγματα για δίθεν υπηρεσίε τη τουρκία στο προσφυγικό όταν μάλιστα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για στήριξη των προσφύγων. δυστυχώ η έκθεση καλωσορίζει την απαράδεκτη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρκίας η οποία καταπατά το διεθνές δίκαιο και θέτει του όρου για εμπόριο ανθρώπων με την τουρκία. η θέση μα είναι ξεκάθαρα η ενταξιακή πορεία της τουρκίας περνά μέσα από τον εκδημοκρατισμό της ίδιας της χώρας αλλά και την υλοποίηση των κυπρογενών της υποχρεώσεων. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αλλά πρώτης, Γόργιος Επιδέος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εάν ένας ε, τρίτος ανεξάρτητος παρατηρητής μπορούσε να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που κάνουμε σήμερα εδώ δεν θα ήξερε τι να καταλάβει. Η Τουρκία παραβιάζει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις εφαρμόζει αυτή. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία της οποίας κατέχει παράνομα τμήμα του εδάφους, απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα αλλά παράλληλα απαιτεί από τις χώρες αυτές να ψηφίσουν για το άγγιγμα των κεφαλαίων της εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες προς την Ελλάδα και η ευρωπαϊκή ένωση την αμείβει με τρία δισεκατομμύρια ευρώ. και επειδή μιλάμε για την ε, έκθεση προόδου της τουρκίας ο ανεξάρτητος παρατηρητής θα μπορούσε να επισημάνει ότι η τουρκία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πρόοδους σε πολύ σοβαρά θέματα παραβίαση του διεθνούς δικαίου παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων φήμωση του τύπου φυλακίσεις όσων εκφράζουν απόψεις που δεν είναι αρεστές στο νέο σουλτάνο της άγκυρας ακριβέστερος βομβαρδισμός των θέσεων των ε, κούρδων μαχητών και στο τέλο, θα κατέληγε στο συμπέρασμα επειδή ακριβώ είναι αμερόληπτο, ότι για να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα μία είναι η λύση άμεση ένταξη της τουρκίας στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Now, on behalf uh, European Commission. Και τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος γιωχάννη Χάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για αυτή την ιδιαίτερως ε, αποκαλυπτική συζήτηση. Ε, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι η Τουρκία είναι ένα στρατηγικό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προκύπτει από τη γεωστρατηγική της θέση, από τον αριθμό των κατοίκων της. Άρα λοιπόν είναι εύλογο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ιδιαίτερο ζωτικό συμφέρον να εξεύρει μια λογική μορφή συνεργασίας. Και ε, βεβαίως σχέση με την Τουρκία έχει τα πάνω και τα κάτω της. Αυτό είναι φυσικό. Αλλά βεβαίως αυτή η μορφή συνεργασίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιεκτική και τα συμφέροντα ε, στη σχέση με την Τουρκία είναι πολύ επίπεδα. Για παράδειγμα, η οικονομική σχέση. Γιατί η Ευρώπη για την Τουρκία είναι ο σημαντικότερος ε, οικονομικός εταίρος και εταίρος για επενδύσεις. Έχουμε 600.000 απασχολούμενους στην Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούνται σε τουρκικές εταιρείες και η Τουρκία είναι για την Ευρώπη ο έκτος κατά σειρά σημαντικότερος οικονομικός εταίρος. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να βρεθεί μια λογική, μια σωστή μορφή συνεργασίας. Επίσης η Τελωνιακή Ένωση είναι ένα σημαντικό μέλημα για μας με το οποίο ασχολούμαι εδώ και έξι χρόνια. Τώρα, η παρούσα κατάσταση με το προσφυγικό έδωσε μια νέα όθηση σε αυτή τη συνεργασία. Αυτό είναι πολύ προφανές και αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράση το οποίο περιλαμβάνει ποικίλα ε, στοιχεία. Η απελευθέρωση της ε, βίζας ε, είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο ήδη έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη στο παρελθόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι το επόμενο βήμα μετά τη θεώρηση εισόδου θα είναι η αυτόματη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, ναι, έχουμε μια εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διεξάγουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ανοιχτή εντολή από το 2005 και έχουμε επιφορτιστεί να διεξάγουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί η εντολή λέει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και εγώ θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να διηγηθούν σε ένα πέρας ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια αξιολόγηση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα άκουσα κατ' επανάληψη πόσο σημαντικό να οι αρχές του κράτους δικαίου στην Τουρκία ε, και πόσο σημαντικό βεβαίως είναι να φροντίσουμε για την εξασφάλισή τους. Κυρίε και κύριοι, μπορώ να πω ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο εφόσον κάνουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μόνο τότε έχουμε έναν μοχλό στα χέρια μας για να κινήσουμε τα πράγματα. Γιατί είναι μια ποιοτική διαφορά το κατά πόσο κάνω ενταξιακές διαπραγματεύσεις ή απλώς ε, προσπαθώ να εντοπίσω κάποια κοινά σημεία με το γείτονά μου. Εμείς ε, ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωση. Ε, έλαβα τις παρατηρήσεις του κ. Λάμπραχτ και άλλων ε, υπόψη μου. Άκουσα με προσοχή τα όσα υπόθηκαν, αλλά θα πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί αντικείμενο της δικής μας εντολής, αλλά το αντικείμενο της εντολής μας είναι να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή και αυτό κατά την άποψή μου μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον εφόσον ε, πραγματικά συσφίξουμε τους δεσμούς της συνεργασίας με την Τουρκία και μόνο τότε μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, το προσφυγικό να επιληθεί με τον προσφυγικό τρόπο. Και με την ευκαιρία αυτή θα μπορούσα να πω ότι το μέσο για την ε, Τουρκία, η διευκόλυνση για την Τουρκία έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή η δήλωση των Τούρκων ότι δεν έχουν δει ούτε ένα σέντς μέχρι στιγμής δεν ευσταθεί. Ε, εμείς ε, βεβαίως χρηματοδοτούμε κάποια προγράμματα στην Τουρκία τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη των εξόδων και τη δημιουργία υποδομών στην Τουρκία για τη στέγαση των προσφύγων στην Τουρκία, ούτως ε, ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική Τουρκία, να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ε, στη χώρα, ούτως ώστε να μπορέσουν άμεσα να επιστρέψουν στη Συρία, εφόσον το επιτρέψει ε, η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα. Εδώ επικεντρώνονται οι προσπάθειές μας, ούτως ώστε τα κονδύλια αυτά να επενδυθούν ε, πρωτίστως ε, σε τέτοιου είδους υποδομές. Ε, με 55 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίσαμε 350.000 άνθρωποι τουλάχιστον μισό χρόνο να έχουν μια στέγαση και ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, με ένα αντίστοιχο ποσό τα παιδιά να μπορέσουν να επισκεφθούν το σχολείο ένα αντίστοιχο διάστημα. Και βεβαίω αυτό συμβάλλει στην ε, βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Γιατί βεβαίω πρόκειται για επικίνδυνο ληστερό έδαφο, αλλά μεταξύ εταίρων είναι αναγκαίο να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και νομίζω ότι αυτό είναι το κοινό μας ενδιαφέρον και το πώς θα διαμορφωθούν ε, τα πράγματα μελλοντικά αυτό θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα εξ του Συμβουλίου η πρώην συναδελφός μας και τώρα Πρόεδρο του Συμβουλίου, η κυρία Χένι Πλάσερ. Έχετε το λόγο σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και ιδιαίτερα επίκαιρη ανταλλαγή απόψεων που καταδεικνύει ότι εμείς από πολλές απόψεις συμμεριζόμαστε και ελπίδες αλλά και ανησυχίες σε σχέση με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συμμερίζονται πολλούς δεσμούς η σχέση μας είναι πολύ παλιότερη από την τωρινή κρίση προσφύγων. Καλύτερη συνεργασία είναι θετική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένα σημείο αναφοράς για την ε, πρόοδο της Τουρκίας στον οικονομικό και πολιτικό χώρο. Όπως ελέγχθη πολλές φορές εμείς δεν συνδέουμε την μετανάστευση με τις συνομιλίες ένταξης. Είναι τελείως χωριστά θέματα. Όπως είπαμε, Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στην περίπτωση της Τουρκίας και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για αρνητικές τάσεις σε ό,τι αφορά τις βασικές ελευθερίες στο κράτο δικαίου και για όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Αν συνεχίσουμε όμως ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις καταστάσεις και την κατάσταση στην Ανατολική Τουρκία με μεγάλη προσοχή και θα εξακολουθήσουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σε όλες τις συναντήσεις και σε όλα τα επίπεδα για το θέμα της φιλελευθεροποίησης των προξενικών θεωρήσεων που ανέφερε ο κύριος Επίτροπος. Ναι, δεν θα κάνουμε κανένα είδος εκτόσεων. Όπως συμφωνήσαμε με την Τουρκία, η απέτηση για βίζα για τους Τούρκους πολίτες μπορεί να αρθεί τον Ιούνιο του 2016 αν εκπληρωθούν όλες οι προδιαγραφές, τα benchmarks. Αν γίνει αυτό πραγματικότητα φυσικά εξαρτάται από την πρόοδο που θα επιτύχει η Τουρκία κάποια ακόμα σχόλια, κύριε Πρόεδρε, για τη συμφωνία της 8ης Μαρτίου. Κατά την άποψή μου αυτή η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό βήμα για να μπορέσουμε να βρούμε μια νόμιμη και ευρωπαϊκή λύση για τα θέματα μετανάστευσης. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, δεν θα είναι πανάκια, αλλά είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, ένα σημαντικό εργαλείο. Όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν επί τη βάση των διεθνών ε, προτύπων και επί τη βάση της αρχής της μη επαναπρόθεσης. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, τα ξέρουμε και δεν θέλουμε να μεταφέρουμε σε άλλους τα προβλήματά μας. Είναι πολύ νωρίς να αξιολογήσει κανείς τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας γιατί η εφαρμογή έχει γίνει μόνο από τις 4 Απριλίου. Να είμαστε σαφείς όμως ότι είναι στο συμφέρον, προς το συμφέρον μας να είναι επιτυχές αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Πλάσερτ. Με αυτό σας αναφέρω ότι έχω λάβει μία σειρά από για την λήξη της συζήτησης και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το επόμενο θέμα τώρα της ημέρας